Ε, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ich erkläre die am 27. November Κηρύττω την ε, επανάληψη της Συνόδου Ολομέλειας που διακόπησε στις 27 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης είναι μια βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Τουρκία είναι μια χώρα υπό